να ανακοινώσω ότι ο κύριος Χουάν Φερνάντε Λόπες Αγγιλά έφυγε από την ομάδα των σοσιαλιστών, των σοσιαλιστών και δημοκρατών και πλέον είναι μη εγκυγραμμένο μέλος από τις 15 Απριλίου και εφεξής. Και θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο